καταδείξουμε τον πλούτο που μπορούν να προσφέρουν οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες της ηλικιακής ε, αυτής ομάδας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία αύριο στις 11.30. Συνεχίζουμε αύριο το πρωί, 3η 13 Σεπτεμβρίου του 2011 στις 9 το πρωί. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.